Sit down, please. Παρακαλώ καθίστε. Cari colleghi. Συνάδελφοι, την περασμένη Παρασκευή 24 Νοεμβρίου επλήγει ένα τζαμί στο, βόρειο, ε, στο Σινά, στη Βόρειο Αίγυπτο. Ε, έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδε